Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την υπομονή σας. Αν θα θέλετε παρακαλώ να κάτσετε. Για να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το σημείο 9, που είναι η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες προτεραιότητες στην πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να σας αναφέρω τι λέει η Επιτροπή στο, στην επιστολή Θέλουμε να κοιτάξουμε ότι είναι προετοιμασμένη η πολιτική για την πνευματική διοκτησία, για την ψηφιακή εποχή και σε ό,τι αφορά τις νέες προτεραιότητες στα επόμενα χρόνια. Η παρουσίαση λοιπόν της δουλειάς που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση θα μας γίνει από την DG για να δούμε τις νέες προτεραιότητες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ευχαριστήσουμε τον ε, υποδιευθυντή για θέματα εσωτερικής αγοράς, επιχειρηματικότητας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος ήλθε να συζητήσει τα θέματα αυτά μαζί μας. Σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που είστε μαζί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνει το λόγο άμεσα μόλις κατέφτασε. Θα έρθουν και τα μέλη της Επιτροπής σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τι σκοπεύουμε σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Ο υποψήφιος ε, Επίτροπος επιμένει λοιπόν και έβαλε σε μεγάλη προτεραιότητα τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και φυσικά το θέμα της ψηφιακής διάστασης. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σημαντικά τα πνευματικά δικαιώματα, το ξέρετε φαντάζομαι, και όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντικά γιατί είναι θέμα ανταγωνιστικότητας. Αν θέλουμε η βιομηχανία μας, ο κλάδος αυτός να συνεχίσει να ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη καινοτομία στην Ελλάδα στην Ευρώπη, συγγνώμη. Και ο καλύτερο τρόπο είναι να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων ε, είναι προσαρμοσμένο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πολλά έχουμε πετύχει λοιπόν με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τη θητεία της. Πολλά πάτυχε λοιπόν η τρέχουσα επιτροπή, αλλά είναι σαφέ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τι νέε προκλήσει και να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο για το μέλλον. Για να βοηθήσουμε τι ε, εταιρείε μα να συνεχίσουν να κάνουν το μουν και στο μέλλον. Ένα βασικό στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο είναι και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ γιατί αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο ποσοστό των επιχειρήσεων στην ε, Ευρώπη και μεγάλο ποσοστό των θέσεων απασχόληση. και είναι επίσης πολύ καινοτόμε. Όπως θα διαπιστώσουμε όμω οι δυσκολίε ε, και ο ρυθμός των πνευματικών δικαιωμάτων ανά μικρομεσαία στην Ευρώπη Είμαστε πίσω στη σχέση με όλο τον κόσμο. Το σύστημα λοιπόν για τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να καταστεί πιο ελκυστικό για τι μικρομεσαίε μα επιχειρήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο επειδή έχουμε τόσε πολλέ μικρομεσαίε, αλλά γιατί θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι μεγάλη πρόκληση λοιπόν για την νέα Επιτροπή και για το νέο Κοινοβούλιο και για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη, γιατί πραγματικά είναι κρίσιμη σημασία. Και πάλι εξετάζοντα αριθμητικά στοιχεία, βλέπουμε ότι σε κάποιε περιπτώσει στην Ευρώπη ε, συγκαζόμαστε και λέμε εντάξει, είμαστε αρκετά καινοτόμοι και δημιουργικοί. Τα αριθμητικά στοιχεία μα διαψεύουν όμω. Έχουμε μείνει πίσω. Για παράδειγμα, το 2018 πάνω από το ίμιση των πνευματικών δικαιωμάτων στον κόσμο ήταν από την Ασία. Και εκείνα τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα που, που ζητά ε, κατοχήρωση πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Η Κίνα είναι πάρα πολύ ενεργή σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στην παρούσα φάση. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μας αντιγράφουν. Όχι, δεν ισχύει αυτό πλέον και να το έχουμε υπόψη μας αυτό αν θέλουμε να αντιτηρήσουμε την εγωνιστικότητά μας. Οι συνάδελφοί μου μου παρουσίασαν, μου προετοιμάσαν ένα μεγάλο κατάλογο το ότι έχουμε πετύχει στο προηγούμενο Κοινοβούλιο και στην προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ ε, εντυπωσιακά όλα αυτά. Δεν πρόκειται να τα αντιτρέξω όλα αυτά. Ζητώ συγγνώμη στους συναδέλφους. Να σας πω ότι κάποια από τα κείμενα τα οποία εγκρίναμε είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά, αν συνδέχει τα εμπορικά ε, μυστικά, σε ό,τι αφορά τι κυβερνοκλοπέ τέτοιων μυστικών, σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των trademarks, σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα πιστοποιητικά προστασία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για κάποιου τομεί, χάρη και στην ε, συνεργασία του Κοινοβουλίου. Και επίση αυτά που κάνουμε για την βιοτεχνολογία και το καθεξή. Αυτό που θέλω να πω για το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε είναι το εξή. Καλή είναι η έγκριση, δεν λέω, αλλά το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά να υλοποιηθούν μεταφέροντας όλα τα στοιχεία αυτά στην εθνική νομοθεσία και εξασφαλίζοντας ότι όλα αυτά πραγματικά λειτουργούν και αναπτύσσονται. Ε, ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα σας ενδιαφέρει, μια νέα φάση αν θέλετε, ένα στοιχείο λοιπόν στο οποίο επιμένω είναι το πακέτο IP το οποίο εγκρίθηκε το 2017 σε ό,τι αφορά το θέμα της υλοποίησης της εφαρμογής. Γιατί πάλι και πάλι όταν μιλάμε για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν στην Ευρώπη, δεν έχει νόημα αν δεν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο. Και από αυτή τη άποψη ε, έχουν γίνει πολλά, αλλά πολλά απομένουν να γίνουν και στο μέλλον. Χαίρομαι που αναφέρω ότι τώρα πια, για παράδειγμα, έχουμε σημαντική πρόεδρο που έχει λάβει η χώρα για το Μνημόνιο Συμφωνίας ε, τα οποία έχουν υπογραφεί και έτσι όλο και πιο πολλοί ε, εμπλεκόμενοι φορείς ε, συμμετέχουν στις ε, συμφωνίες αυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν θέλουμε να είναι σωστή η υλοποίηση και εφαρμογή τη προστασία των δικαιωμάτων γενετική ιδιοκτησία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι βασικοί φορεί, οι βασικοί παράγοντε του οικονομικού κόσμου συμμετέχουν και εξασφαλίζουν και προσπαθούν να εφαρμόσουν τα δικαιώματα γενετική ιδιοκτησία. Από αυτέ τι άποψει, λοιπόν, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι περήφανοι για αυτά που πέτυχαν. Γιατί πέρσι ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό ο αριθμό των κειμένων που ε, εγκρίθηκαν, ο αριθμό των προτάσεων που εγκρίθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, ε, πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουμε πετύχει, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί και στο μέλλον. Πώ θα δημορφωθούν τα πράγματα στα πλαίσια τη νέα επιτροπή. Τώρα να κάνω και μια σημαντική σημείωση. Δεν είμαι, κυρία Γκουλάρ, και δεν ξέρω τι θα έρθει να σας πει. Δεν είμαι σε καμία θέση να προκαταλάβω αυτά που θα σας πει. Εδώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Όπως και να έχει όμως, θα ήθελα να σας δώσω μια γεύση του τι συζητάμε στο δικό μου επίπεδο, χωρίς να μπορώ φυσικά να προβλέψω τι πρόκειται να δηλώσω στην επόμενη εβδομάδα στις ακροάσεις και όταν θα σας επισκέπτεται πιο τακτικά. Καταρχάς, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σε ό,τι αφορά την ενιαία πατέντα. Ακόμα λοιπόν είναι προσυζήτηση σε ό,τι αφορά το θέμα του κώδικα και το σχετικό δικαστήριο. Θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν σύντομα. Έρχομαι σε πολλές διαφορετικές ε, θητείε έχω έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο για να εξηγώ τα ίδια πράγματα. Είναι σαφέ ότι το τρέχον σύστημα είναι πολύ περίπλοκο, ιδιαίτερα για τι επιχειρήσει μα και είναι πάρα πολύ ακριβό και για τι μικρομεσαίε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει το σύστημα αυτό, το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνία, θα πρέπει να καταστεί πιο λειτουργικό, πιο απλό και λιγότερο ακριβό. Αυτό πραγματικά το χρειαζόμαστε αν θέλουμε να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία και την ανάπτυξη γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο. Δεύτερο στοιχείο. επίσης. Ε, ε, ολοκληρώνουμε την αξιολόγησή μας σε ό,τι αφορά το τρέχον ε, ευρωπαϊκό σύστημα για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασία σε ό,τι αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ξέρουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, Πολλέ συζητήσει έχουν γίνει ήδη για το θέμα αυτό. Αλλά είναι σαφές ότι αν υπάρχει μια πιο ενιαία προσέγγιση και μια μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, είναι εντυπωτικό. Και πάλι βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγηση. Δεν μπορώ να προκαταβάλω και να προβλέψω οποιαδήποτε απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτό προφανώ θα πρέπει να το κοιτάξουμε γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το μέλλον του φαρμακευτικού κλάδου. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με το βασικό θεμελιώδε δικαίωμα του πολίτη να έχει πρόσβαση στα σωστά φάρμακα. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό και το εξετάζουμε. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι και η θέση του Κοινοβουλίου. Μία άλλη αξιολόγηση που λαμβάνει η χώρα είναι η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων. Εξετάζουμε λοιπόν το τρέχον σύστημα, το αξιολογούμε και προσφάτως ε, κάναμε μία δημόσια διαβούλευση από αυτό. Το βασικό μήνυμα που πήραμε από τη διαβούλευση είναι το εξή, ότι καταρχά το σύστημα λειτουργεί αρκετά καλά, δεν είναι κακό, αλλά προφανώ θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα νέα σχέδια και πρότυπα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύονται, να λάβουμε υπόψη επίση τι νέε τεχνολογικέ εξέλιξει που έχουν λάβει η χώρα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το 3D printing, τρισδιάστατη εκτύπωση. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα αυτό. Έχει γίνει και ε, μια, ένα ψήφισμα για το πνευματικά δικαιώματα και την ταιριαστή εκτύπωση. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στα τέλη του χρόνου. Είναι προφανώ ένα καυτό θέμα. Και χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε απλά να το αφήσουμε. Είμαι υπεύθυνο και για θέματα ε, διαστήματο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, νέα συστήματα για τις, ε, τα συστήματα διαστημικά και πολλά από αυτά εκτυπώνονται σε τριδιαστατό επίπεδο. Να σας ε, μιλήσω επίσης για κάποια θέματα τέτοια. Όλοι τα συζητάμε ε, φυσικά τα θέματα αυτά. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαφές ότι έχει καταστεί όλο και πιο βασικό στοιχείο και στις πραγματικότητάς μας η τεχνητή νοημοσύνη, στην οικονομία μας, στις εξελίξεις κτλ. Είναι σαφέ ότι το θέμα αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και προφανώ από πλευρά πνευματικών δικαιωμάτων επίση είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε από την άποψη αυτή. Για έναν απλό λόγο και πάλι. Γιατί όταν μιλάμε για πνευματική, για τεχνητή νοημοσύνη, δεν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που το συζητάμε αυτό. Και σε άλλα μέρη γίνεται ε, μεγάλες επενδύσεις στην Κίνα, στη ΣΥΠΑ. Αν δεν θέλουμε λοιπόν και πάλι να μείνουμε πίσω, τελευταία και καταδεδομένη, θα πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα αυτά τα θέματα. Τελευταίο λοιπόν θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο, πρέπει να το εξετάσουμε από πλευρά πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί ανακύπτουν και ζητήματα ηθικά, δεντολογικά. Για να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Μία, ένα μηχάνημα μπορεί να θεωρηθεί ως εφευρέτης. Εύκολη ερώτηση, απλή. Η απάντηση όμως είναι πολύ δύσκολη. Τέτοιου είδους ζητήματα καλούμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε. Και για να είμαστε να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Δεν νομίζω ότι η κυρία Γκουλάρ την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε θέση να δώσει μια οριστική απάντηση, γιατί είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα αυτά. Αλλά το ότι είναι περίπλοκα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να τα εξετάζουμε. Δεν θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να σκεφτούμε ποιε θα είναι οι συνέπειε από τι άποψει αυτή, λοιπόν ο διάλογο με το Κοινοβούλιο είναι ουσιώδος σημασία και με του υπόλοιπου φυσικά φορεί, αλλά το, το Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούν να μπουν όλα αυτά στους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μία πτυχή που είναι πολύ σημαντική, το ανέφερα και αρχικά και θα πρέπει να το εξετάσουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι καινοτόμες μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν αρκετά τα δικαιώματα πραγματικής δικτυσίας στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό αυτό και βλέπουμε ότι στην Ευρώπη μόνο 9% των ευρωπαϊκών ε, μικρομεσαίων. 9%. Ένα είδους ε, δικαίωμα διανεκτικής ιδιοκτησίας. Μόνο 9% κοιτώντα ε, τι γίνεται στι μεγάλε επιχειρήσει, 36% είναι το αντίστοιχο ποσοστό. Και κοιτώντα τι γίνεται στη ΗΠΑ, επίση είναι πολύ πιο ψηλά τα ποσοστά από ό,τι στην Ευρώπη. Μεγάλο λοιπόν και πραγματικό το πρόβλημα. Φυσικά αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένου λόγου. Είναι ακριβά τα δικαιώματα δεν είναι ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολη διαχείρισή του. Αλλά αυτέ οι εξηγήσει δεν μα ικανοποιούν γιατί Επαναλαμβάνω ότι σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο με τόσε πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι δικέ μα δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το IPR, τα δικαιώματα ειδική ιδιοκτησία. Υποτίθεται ότι προωθούν την καινοτομία. Αν δεν τι χρησιμοποιούν λοιπόν οι εταιρείε μα, έχουμε πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά μπορούμε να απλοποιήσουμε το σύστημα IPR, αλλά δεν είναι απλό. Όπω ξέρετε λοιπόν, τρέχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να δούμε μαζί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς μπορούν να, βελτιώσουμε το σύστημα IPR. Οργανώνουμε επίσης 14 Νοεμβρίου με την Επιτροπή των Περιφερειών και με την Φιλανδική Προεδρία ένα μεγάλο, μια μεγάλη εκδήλωση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε λοιπόν τι ιδέες υπάρχουν. Και πάλι πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι θεμελιώδου σημασία για την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε πόσο σημαντικέ είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για την ε, οικονομία μα και να μην λύσουμε το θέμα αυτό. Αν δεν βρούμε μια σωστή λύση, και φυσικά δεν πρόκειται να υπάρξει μια μαγική λύση, θα πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμό λύσεων. Αν δεν είμαστε σε θέση λοιπόν να βρούμε μια λύση για το πρόβλημα αυτό, πολύ απλά θα μείνουν πίσω οι επιχειρήσεις μας και θα φταίμε εμείς και στη τελική ανάλυση αυτό τι σημαίνει ότι θα χαθούν θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτό πολύ απλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πολύ δύσκολο λοιπόν το θέμα αυτό. Περίπλοκο. Και φυσικά δεν είναι όλε οι μικρομεσαίε ίδιε. Οι μικρομεσαίε στο Βέλγιο δεν είναι ίδιε με αυτέ τη Γερμανία. Αλλά και πάλι το πρόβλημα είναι πραγματικό. Θα πρέπει να το επιλύσουμε. Τέλο, τελευταίο σημείο όπου πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε απομονωμένοι. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή και το θέμα λοιπόν τη ε, παγκόσμια σύγκληση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα δυνητική ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε αυτό λοιπόν στην Ευρώπη. Σε κάποιε περιπτώσει οι επιχειρήσει χάνουν τα δικαιώματά του όταν βγαίνουν εκτό Ευρώπη. Και αυτό φυσικά δρά ανασφαλτικά. Δεν τολμούν να βγουν εκτό Ευρώπη γιατί, γιατί τα προγράμματα δεν είναι. Ε, ε, προστατεύουν αρκετά, δεν είναι σωστά στην προστασία. Αλλά και πάλι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία. Στις επιστολέ Αποστολή τη κ. Φαντελέιεν τονίζεται αυτό ο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο παγκόσμιο προσκήνιο. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτούν αυτέ οι εταιρείε και εκτό Ευρώπη. Γιατί, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρχει και εκτό Ευρώπη τέτοια ανάπτυξη. Είναι μεγάλη πρόκληση, προφανώ. Αλλά αυτά τα θέματα καλούμαστε να τα συζητήσουμε. Άρα, νομίζω ότι σας παρέθεσα και σας παρουσίασα πολλές προκλήσεις. Αλλά ξέρουμε ότι αν δεν συνεργαστούμε για να επιλύσουμε τα θέματα αυτά, για να βρούμε λύσεις, το επόμενο κοινοβούλιο σε πέντε χρόνια δεν θα είναι σε καλύτερη θέση για να επιλύσει τα θέματα αυτά. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αναζητούμε λύσεις οι οποίε θα είναι δύσκολες, δυσέβρετε, δεν θα είναι εύκολε στην εφαρμογή, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ιδάλω σε 5, 10, 15 χρόνια δεν θα είμαστε σε καλύτερη θέση. Δεν έχω λοιπόν συγκεκριμένε λύσει να προσφέρω, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει η συζήτηση μαζί σα για να δούμε πού θα βρεθούμε στο τέλο τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε τις προτεραιότητες σας κύριε Ντελσό. Ο κύριος Μπρέγια τότε και μετά τα υπόλοιπη. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, πρέπει να δούμε πιο διαφοροποιημένα και πιο ρεαλιστικά την πνευματική ιδιοκτησία και τα σχετικά δικαιώματα η αύξηση της καινοτομία ε, είναι θετική, αλλά οικονομικά μετά από κάποιο επίπεδο πέραν της κάποιου βαθμού καινοτομία και ε, ανάπτυξης θα πρέπει να έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα διπλώματα την χάνουν κατάχρησης. Να σας περιγράψω τι γίνεται στη Γερμανία όπου η οδηγία εφαρμογής των δικαιωμάτων ε, πνευματική ιδιοκτησίας οδηγεί τι επι, ε, να μην ε, μπορούν να ανοίξουν δίκτυα Wi-Fi χωρίς ολόκληρη διαδικασία, χωρίς να πληρώνουν για την προστασία των ε, password, για παράδειγμα. Κάτι που επιβαρύνει την οικονομία μας. Ας έχουμε λοιπόν μια προσέγγιση κάπως πιο διαφοροποιημένη. Δεύτερον, γιατί δεν χρησιμοποιούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καινοτόμε ε, και προωθημένες επιχειρήσεις. Διότι η απάντηση για μένα είναι απλή. Δεν έχουν όρεξη να τρέχουν σε δικαστήρια, θέλουν να κάνουν δουλειά. Προτιμούν λοιπόν να μην χρησιμοποιούν τέτοια δικαιώματα γιατί θέλουν να προστατεύουν την καινοτομία τους με άλλο τρόπο ή ε, βρίσκουν άλλους τρόπους γενικότερα. Καλύτερα να προστατεύει, βρίσκουν άλλους τρόπους να προστατεύουν την καινοτομία τους και όχι τα νομικά, το νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, αν επιχειρήσει αποφασίζουν να μην προστατεύουν την καινοτομία τους με δικαιώματα, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε κι εμείς. Άλλοι συνάδελφοι και μετά θα επανέλθουμε για σχόλια. Κύριε και μετά ο κύριος Στανκιανέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και την παρουσίασή σας. Ε, θα ήθελα καταρχάς να σας ενθαρρύνω να συνεχίζετε να δείχνετε τέτοιο επίπεδο φιλοδοξίας και να συζητάτε τέτοιε ιδέε μαζί μα, γιατί έχω και την αίσθηση ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη και όλο και πιο πολύ καθίσταται επίγον το θέμα αυτό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όλα αυτά τα θέματα και να δούμε πώ η Ευρώπη μπορεί με ενιαίο τρόπο να προσπιστεί τα συμφέροντά της. Γιατί το διαπιστώσαμε και στην προηγούμενη θητεία, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να προασπίζονται πιο πολύ τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Δεν προσπαθούν τόσο πολύ να συνενώσουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ευχαριστήσω που είσαστε τόσο φιλόδοξοι και να σας καλέσω να συνεχίσετε να δείχνετε τέτοιο επίπεδο φιλοδοξίας και κυρίως ε, από πλευράς ΕΛΚ και από την πλευρά της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων θα σας ε, υποστηρίξουμε σε αυτή την υψηλή φιλοδοξία σας γιατί πολύ απλά έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει στα βήματα αυτά που καλούμαστε να πάρουμε. Όπως σας είπα, το θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος Μπράιερ, του πού βρισκόμαστε, τι ισορροπίες πρέπει να πετύχουμε για να έχουμε αυτό που επιθυμούμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε και ε, τα ενιαία ευρωπαϊκά συμφέροντα τα οποία να υποστηρίζονται. Από την άλλη, να μην καταστρέψουμε και τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Πώς μπορούμε να πετύχουμε το γεγονός ότι θα σταματήσει η πώληση διπλωμάτων ευρύς συνταχνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις πτυχές αυτές που αναφέρατε, τεχνητή νοημοσύνη, τρίτη διαφορετική τύπωση, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ουσιώδη. Σας καλώ λοιπόν να συνεχίσετε τις προσπάθειες και θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι σε αυτούς τους τομείς όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται με λυγκιώδους ρυθμούς θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλη ταχύτητα στην ανταπόκριση, την νομική. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε πολύ γρήγορα να εργαστούμε για να μπορέσουμε επίσης και να διορθώνουμε πιο γρήγορα όπου γίνονται σφάλματα. Να υπάρχει ένα σύστημα λοιπόν έκτακτης ε, ανταπόκρισης, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε και να προσπαθούμε εκ των προτέρων να ξεκαθαρίζουμε την ε, κάθε αντιπολεπτομέρεια. Θα πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι και να προσπαθούμε να επιλύουμε προβλήματα όπου αυτά παρουσιάζονται. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και θα πάρει το λόγο ο κ. Βόλκερ και μετά το λόγο θα έχει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ο κ. Βόλκερ να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή και χαίρομαι που μπορούμε να συνεργαστούμε εκ νέου. Είναι πολύ φιλόδοξη η ατζέντα που μας παρουσιάσατε σήμερα. Είπατε ότι φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και η Επίτροπος για τα θέματα αυτά. Βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας. Χαίρομαι που το SPC ξαναμπήκε στην ημερήσια διάταξη για έναν ε, επιπλέον τομέα εφαρμογή από ότι σε σχέση με την προηγούμενη θητεία. Νομίζω ότι καταφέραμε να συμπληρώσουμε μια καλή πρόταση στην προηγούμενη θητεία και νομίζω ότι στην όλη συζήτηση άκουσα ότι κυρίως πρόκειται για θέματα που αφορούν την οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό στέκει. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι στα δικαιώματα γενετικής ιδιοκτησίας τρύφεται και μια κοινωνική λειτουργία, γιατί αυτός που εφευρίσκει κάτι προφανώς και έχει δικαίωμα, αλλά και η κοινωνία έχει δικαίωμα να ωφεληθεί από την εφεύρεση την κάθε εφεύρεση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι μου φαίνεται ότι θα παρουσιάζεται όλα πιο πολύ από την οπτική γωνία της οικονομίας σε ό,τι αφορά τον εφευρέτη. Όλοι συμφωνούμε ότι χωρίς ε, χωρί δημιούργημα δεν μπορεί να υπάρξει δημιουργία. Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να δημιουργήσει ένα μηχάνημα, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό θα έχουμε ακόμα χρόνο. Ένα ακόμη ομιλητή. Έχουμε στον κατάλογο να ακούσουμε τον κύριο Ντεμπλάνκο πρώτα και μετά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για την ε, ομιλία σας. Σημειώνω και πόσο ευγενικά είπατε ότι εσείς μπορείτε να απαντήσετε σε να λαγούν στη θέση σας, αλλά εσείς είστε διευθυντής. Επομένως, ε, σίγουρα απαντάτε στο επίπεδο του διευθυντή και όχι του επιτρόπου. Εγώ θέλω να θέσω μία απλή ερώτηση. Δεν θεωρείτε, και συμφωνώ με όσα είπατε, δεν θεωρείτε ότι ένα σημαντικός αγώνας κατά της παραποίησης αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία της διανοητικής διοκτησίας. και αναφέρομαι στις ε, αρμοδιότητές σας ε, ως διευθυντής. Ε, μπορείτε να μας απαντήσετε ποιες δράσεις μπορούμε να φανταστούμε για το μέλλον. Δεν ε, αναφέρομαι όσα έχουν γίνει ήδη, γιατί η παραποίηση καταπολεμείται έχοντα κατά νου ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από, λείπουν από τις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις που κάνουν θυσίες, κάνουν έρευνα, επενδύουν και κατόπιν βλέπουν αυτό που βλέπουμε και θα μιλήσω για την Ιταλία, αλλά πιστεύω ότι και αλλού το βλέπουμε αυτό, ότι υπάρχει μια μεγάλη αγορά παραποίησης που συχνά γονατίζει ολοκληρές κοινότητες. που βασίζονται στην εφευρετικότητά τους. Σας ευχαριστώ για τα όσα μπορείτε να μας πείτε. Έναν ακόμα μιλητή έχουμε, λυπάμαι. Ο κ. Δεμπλάνκο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Όμως μου έλειψε κάποια περαιτέρω αναφορά στο δίκαιο της διανοητικής διοκτησίας και στο δικαίωμα του δημιουργού. Σε ό,τι αφορά και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Και μου έλειψε ε, και το να μας σχολιάσετε ποιες είναι οι προοπτικές που έχει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά και τα όσα λέγονται στην τελευταία οδηγία για το copyright. Και επίσης, ε, αν θα υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ό,τι αφορά το δικαίωμα του δημιουργού, το δικαίωμα στην αμοιβή, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και μια σκέψη. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποχρώσεις ε, στην ιδιωτική διοκτησία. Στην ισπανική νομοθεσία θεσπίζεται ε, ότι θα πρέπει να ακολουθούν οι νόμοι ε, και το τι ισχύει στο κοινωνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο νομικό που να είναι ελεύθερο στην ερμηνεία. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούμε στην Ευρώπη για ιστορικούς ε, και γεωγραφικούς λόγους, αλλά και προκειμένου να εξεχρονίσουμε την οικονομία μας σε παγκοσμίο επίπεδο. Δεν είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί σε πολλά πράγματα, ε, όπου πρώτα είχαμε ανταγωνισμό. Ο μόνος ε, τρόπος που μπορούμε να δημιουργήσουμε πόρους από το τίποτα είναι η δημιουργικότητα πρακτικά. Και ε, πρέπει να ε, υπάρχει ουσιαστικά το δίκαιωμα στην προστασία της νοητικής διοκτησίας, αλλά πρέπει να δούμε ε, ουσιαστικά και το πώς η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας σε ερωτήσεις που σας έθεσα. Ευχαριστώ. Έχω ένα σχόλιο κι εγώ και κατόπιν θα σας δώσω το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που δώσατε έμφαση στις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός τομέας και πρέπει να το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιόμουν αν ε, έχετε ε, σκεφτεί να ε, υποστήριξετε τις γυναίκες που είναι επικεφαλής τέτοιων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο. Ξέρω ότι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν διευθυντές γυναίκες ε, και πολλές φορές δεν νιώθουν ε, ότι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον κόσμο της τεχνολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να, να μου πείτε αν αυτή η πτυχή έχει ενταχθεί στο μελλοντικό σας έργο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ε, και εμεί ζητάτε συγγνώμη, ότι έχετε τόσες ερωτήσεις δείχνει ότι ενδιαφέρεστε. Εγώ το βλέπω θετικό αυτό. Και επίσης σας ευχαριστώ για την ευρεία υποστήριξή σας. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σημεία Όπω είπατε δεν έχουμε ύλε ε, στην Ευρώπη, Α είμαστε σαφεί. Έχουμε πολύ περιορισμένο αριθμό πρώτων υλών. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσει απασχόληση για τα παιδιά και τα εγγόνια μα, ε, έχουμε την δημιουργικότητα και την κοινοτομία ω περιουσιακό μα στοιχείο. Αν δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με την κοινοτομία μα, γιατί δεν έχουμε φυσικού πόρου στην Ευρώπη, τότε θα μείνουμε πίσω σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Καινοτομία λοιπόν και η ικανότητα να εφεύρουμε νέε λύσει είναι κάτι θεμελιώδε για όλου εμά του Ευρωπαίου. Το πρώτο στοιχείο ήταν αυτό. Δεύτερο, αυτή η συζήτηση για το γεγονό ότι τα δικαιώματα εκκλησία είναι περιορισμό και θα μπορούσε να υπάρχουν καταχρήσει, ε, ναι, ισχύει. Σε ορισμένε περιπτώσει έχουμε καταχρήσει ε, των IPR και δώσω ορισμένα παραδείγματα που μάλλον πήγαν πολύ μακριά. Όμως ε, δεν έχουμε βρει τίποτα καλύτερο από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αν δεν μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά θα εφαρμόζονται στην Ευρώπη, τότε τι θα γίνει η καινοτομία, ε, τότε θα κατοχυρηθεί από κινέζικες εταιρείε που θα χρησιμοποιούν τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως, δεν είναι θέμα να αγωνιστούμε κατά των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να θεσπίσουμε ένα μηχανισμό ώστε να μην υπάρχουν καταχρήσεις των δικαιωμάτων. Σίγουρα πρέπει να το διερευνήσουμε αυτό, αλλά είμαστε σαφές. Σαν ε, δεν ε, είναι οι εταιρείε μας που θα καταχωρούν ε, δικαιώματα, τότε θα είναι κάποιοι άλλοι. Και φυσικά το ωφέλη θα πάνε σε κάποιον άλλο και όχι στις ευρωπαϊκές εταιρείε. Έτσι λοιπόν, από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να συνεχίσουμε με την εφαρμογή και θα πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε υπερβολικά δικαιώματα. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θέλω να επιμείνω και νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι το εξή. Αν δείτε τι μελέτε, όλε οι ΜΜΕ που έχουν ε, περισσότερα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία ε, έχουν καλύτερου μισθού και είναι πιο παραγωγικέ. Έτσι λοιπόν, το να μπορεί ω ε, μικρομεσαία εταιρεία να είσαι σε θέση να έχεις δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας σε βοηθούν να είσαι πιο παραγωγικός και να πληρώνεις καλύτερους μισθούς, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι λοιπόν κάτι ίσονο σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα φυσικά όταν μιλάμε για τα δικαιώματα πνευματικής δικτύας και είπατε το θέμα της εφαρμογής είναι σημαντικότατο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ε, ότι έχουμε ορθή εφαρμογή. Και να πω ότι όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δεν ε, ε, πρέπει μόνο η Κομισιόν να κάνει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει και οι εθνικέ αρχέ να είναι πιο αποτελεσματικέ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ενισχύσουμε του δεσμού συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και να χρησιμοποιούνται και οι φυστάμενε βάσει δεδομένων στα κράτη-μέλη αν ε, δεν δημιουργήσουμε αυτή το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ όλων των ε, ε, αρχών, τότε θα έχουμε παραποίηση και θα χάσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και μία όθηση όπου όλα τα κράτη-μέλη θα δεκτούν να συνεργαστούν πλήρως και να θεσπίσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις, τα δικαιώματα πνευματικής διεκτησίας, γιατί όπως είπατε η παραποίηση του ζημιώνει όλους. Τώρα, για το copyright. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και φυσικά υπό το προηγούμενο κοινοβούλιο είχαμε πολύ δύσκολες συζητήσεις για να βρούμε συμβιβασμό. Και πάλι δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Νέας Επιτρόπου, δεν είμαι ένα επίτροπος, ε, όμως ε, ανοίγουμε την συζήτηση ε, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ε, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που έχουν ε, συμφωνηθεί και επίσης είναι σημαντικό να δούμε το μέλλον και να συζητήσουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να δούμε τι έχει συμφωνηθεί καταρχήν, πώς θα το εφαρμόσουμε και να δημιουργήσουμε, συγγνώμη, να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Και ξέρουμε ότι στα κράτη-μέλη ε, και ο κλάδος συζητά για πιθανές κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα, για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ε, των μηχανών, ε, κοιτάξτε, ήμουν κάπως προκλητικός όταν έθεσα την ερώτηση. Όμως, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε ότι έρχεται και θα τεθεί επιτάπητο στο ζήτημα και θα πρέπει να το προλάβουμε. Τώρα, για τις γυναίκες διευθυντές είναι ένα ευρύτερο θέμα, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη γενική μας διεύθυνση. Εξετάζουμε και τη στρατηγική για τις ΜΜΕ, γιατί είναι και μέρος της επιστολής της Νέας Προέδρου και το θέμα της γυναικείας διοίκησης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενημερωτικά. Δεν ε, μιλώ για τις ΜΜΕ, αλλά στις μεγάλες εταιρείες όπου έχουμε ε, πολλές γυναίκες στο δικό συμβούλιο βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μία μελέτη το έχει αποδείξει αυτό, όμως οι γυναίκες επιχειρηματίες και ο ρόλος της ΜΜΕ είναι ένα ευρύτερο θέμα. Είναι πολύ πιο ευρύ από τα θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι συνολικά απάντησα σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και φυσικά θα δούμε προς το που θα οδεύσει η νέα Κομισιόν. Έχω μία ακόμα ερώτηση. Ποιο Βόλκαν έχει, νομίζω ότι αυτό προέρχεται από τις ε, ερωτήσεις σας. Μια γρήγορη ερώτηση. Μιλήσατε για τις επόμενες συζητήσεις για το φάκελο του, των copyright και την συνάντηση με τους εμπλεκόμενους που θα οργανώσει η Επιτροπή. Έχετε στοιχεία για το πόσοι ενδιαφερόμενοι θα μετάσχουν σε αυτή την συνάντηση, σε αυτό το διάλογο και αν ναι, μπορείτε να μας πείτε πόσες μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σύνδεσμοι θα μετάσχουν. Ξέρω ότι είναι αυθόρμητη η ερώτηση. Αν έχετε όμως κάποια σχετικά στοιχεία θα ήταν πολύ θετικό. Πολύ. Δεν έχω τα ακριβή στοιχεία. Αλλά αν θέλετε προτείνω να έρθουμε με συγκεκριμένα στοιχεία ανακατηγορία επιχειρήσεων κλπ. Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα που δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω θα είναι πολύ θετικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ να ανταλλάσσουμε απόψεις. Ήταν καλό που ακούσαμε τις ε, φιλοδοξίες σας για την επερχόμενη επιτροπή. Αυτό είναι το τελευταίο θέμα στην επιτροπή μας για σήμερα. Άτυπα σας λέω ότι έφυγαν δύο προσκλήσεις. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Αν θέλετε περισσότερα σε προσωπικό επίπεδο μετά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ που κάτσετε μέχρι τώρα εδώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.